κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα καλωσορίσω και στη σημερινή συνεδρία τη Επιτροπή μα. Θα σα ζητήσω συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά όπω ξέρετε, περιμένουμε πάντω του συναδέλφου οι οποίοι βρίσκονται σε άλλε συνεδριάσει και πρέπει να είναι εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω του εκπροσώπου όλων των διπλωματικών αποστολών και του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τον κύριο Νταλαρίτσια, προϊστάμενο τη Διεύθυνση για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική, τον κύριο Κωνσταντίνο Βέρδο από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνού Συνεργασία και Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Να σα πω ότι η διερμηνία παρέχεται στην Αγγλική, Ισπανική, Ελληνική και Ιταλική και η παθητική θα είναι η Γαλλική. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Το σχέδιο της μερίσιας διάταξης έχει διανεμηθεί στα αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρηθεί ότι η μερίσια διάταξη έχει εγκριθεί. Τα πρακτικά της συνεδρίας της 27 Απριλίου του 2017 περιλαμβάνονται στο φάκελο και αν δεν υποβληθούν τροποποιήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας θα εγκριθούν χωρίς αλλαγή ή αν γίνουν κάποιες αλλαγές θα συμπεριληφθούν και αυτές. Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω στα μέλη ότι η αντιπροσωπεία είχε προγραμματίσει επίσκεψη στην Κούβα για την εβδομάδα από τις 30 Οκτωβρίου και στις 3 ε, Νοεμβρίου του 2017. Όπως θυμάστε είχαμε λάβει προφορική επιβεβαίωση από τις κουβανικές αρχές για την πρόθεσή τους να μας δεχθούν. Δυστυχώς όμως, λόγω της μεγάλης καταστροφής που προκάλεσε ο τυφώνας Σύρμα, το νησί στο νησί, η αυτού εξοχότητα πρέσβυρα η κυρία Κοϊκοτσέα, με ενημέρωσε γραπτό στι 14 Σεπτεμβρίου του 2017 ότι η επίσκεψη της αντιπροσωπείας δεν ήταν εφικτή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το ηλεκτρονικό μήνυμα σας επισυνάπτεται στο φάκελο και θέλω να διαβεβαιώσω τα μέλη ότι από την πλευρά μου θα εργαστώ ώστε να πραγματοποιηθεί μια αντχόκα επίσκεψη τη αντιπροσωπεία στην Κούβα σε μεταγενέστερη ημερομηνία κατά το επόμενο έτος. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία μα σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ικαράγουα και το Ελ Σαλβαδόρ κατά την 7η εβδομάδα από τι 12 έω 16 Φεβρουαρίου του 2018. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με τι επισκέψει των αντιπροσωπιών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τι λεπτομέρειε τη επίσκεψη κατά την επόμενη συνεδρία τη αντιπροσωπείας. Περνώντας σε ένα άλλο θέμα, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η κυρία Λολίτα Τσαβέθ, Ιξκακουίκ, υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Γουατεμάλα, είναι μεταξύ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροβ 17. Είναι μέλος του Συμβουλίου των Λαών του ΚΙΤΣΕ, οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία των φυσικών πόρων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την χωρίς όρια και κανόνες εκμετάλλευση της μεταλλουργίας, της υλοτομίας, των υδροηλεκτρικών και γεωργιομηχανικών τομέων στην περιοχή. Η κυρία Ιξκακουίκ έχει υποστεί πολυάριθμες απειλέ και είχα χαρά να τη συναντήσω, αυτή τη χαρισματική γυναίκα, κατά την τελευταία συνεδρία της στο Στρασβούργο. Όπω γνωρίζετε, η διάσκεψη των Προέδρων, η αρχηγή των πολιτικών ομάδων και ο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επιλέξει την προσωπικότητα στην οποία θα απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάροβ για το 2017 μεταξύ των τελικών υποψηφίων στι 26 Οκτωβρίου. Περνώντα ένα άλλο ζήτημα, θέλω να σα ενημερώσω ότι η ύπατη εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μονκερίνη, όρισε την κυρία Μαρίζα Ματία, Ευρωβουλευτή τη GUNCL από την Πορτογαλία, ως επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών στην Ονδούρα. Θα ήθελα να συγχαρώ, να συγχαρώ την κυρία Ματίας και να υπενθυμίσω ότι οι γενικές εκλογές στην Ονδούρα θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου του 2017. Η αντιπροσωπεία μας θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα αποτελέσματα της αποστολής στην επόμενη συνεδρίασή τη. Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι έλαβα σημείωμα από την πρεσβεία της Ονδούρα με το οποίο μας ενημερώνει σχετικά με την απόφαση του οίκου για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ονδούρας από Β1 έως Β2. Πρόκειται για μια ευχάριστη είδηση που δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώνεται. Εγώ απλά να πω στο σημείο αυτό ότι περιμένουμε να δούμε τη βελτίωση αυτή να μεταφράζεται στην απτή μείωση της στόχιας, της ακραίας στόχιας και των ανισοτήτων. Στην έκθεση που θα συζητήσουμε σήμερα επιβεβαιώνεται ότι τέτοια μείωση από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει. Το σημείωμα επισυνάπτεται στο φάκελο για τα μέλη. Σχετικά τώρα με την ολοκλήρωση της αποστολής της Επιτροπής Ανάπτυξης στην Ονδούρα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως και στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017. Ο σκοπό τη αποστολή τη Επιτροπή τη ΔΕΒΕ στην Ονδούρα ήταν να εξετάσει εάν τα προγράμματα που υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ικανοποιητικά, κατά τρόπο επικοδομητικό σε μια σειρά από Τα μέλη τη αντιπροσωπεία προέβησαν σε λεπτομερή έλεγχο των προγραμμάτων σε τομεί όπω η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου, η ενίσχυση των θεσμών, η κοινωνική ισότητα και η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι και η δική μα αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ονδούρα από 18 έω 20 Φεβρουαρίου του 2015 και με την ευκαιρία αυτή προέβη επίση σε λεπτομερή έλεγχο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντο και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν εκ νέου για την κατάσταση στη χώρα, να συγκρίνουν την κατάσταση και να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, την κυρία Σάντζεθ, Λόλα Σάντζεθ, η οποία συμφώνησε να ενημερώσει την αντιπροσωπεία μας για τα ευρήματα της αποστολής λίγο μετά την επίσκεψη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, που μαζί με την επικεφαλής της αντιπροσωπείας κυρία Σάντζεθ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε στα χέρια μας την πλήρη έκθεση της αποστολής της ΔΕΒΕ για τη συνεδρίαση αυτή. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Σάντσεθ, Ευρωβουλευτή της Γκουέντζιέλ, επικεφαλή της αποστολής της Σχετικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη στην Ονδούρα και να μας, ε, για την, να μας ενημερώσει σχετικά με το όσα ε, εκεί είδαν και συζήτησαν. Κυρία Σάντσεθ, έχετε το λόγο. Muchas gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ονδούρα είναι η πιο φτωχή χώρα της ε, ε, Λατινικής Αμερικής ε, αλλά με πληθυσμό πάνω από 8 εκατομμύριο θεωρείται μια ε, χώρα μεσαίου εισοδήματο. Ε, για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη και έχουμε και πολύ περιορισμένο αριθμό γεωργικών προϊόντων και ένα τομέα κλωστοϊφαντοργίας στον οποίο οι συνθήκες εργασίας αποτελούν λόγο πολύ σοβαρής ανησυχίας. Ε, Πράξει, βίε, απειλέ, οργανωμένο εγκλήματα και οργανωμένη ατιμορρησία επίσης υπάρχει. Ε, η Ονδούρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά δολοφονιών ανά τον κόσμο. Η ε, φτώχεια επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια και υπήρχε και ένα πολύ σημαντικό ε, πρόβλημα δολοφονιών ε, ε, ακτιβιστών για θέματα περιβάλλοντος. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι ο Κάθερες. Στην περιοχή είναι η πιο φτωχή χώρα μετά από τη Βολιβία. Ο λόγο τη επίσκεψη τη επιτροπή ε, στην Ονδούρα ήταν να δούμε πώ εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα δημοκρατία, κράτου δικαίου, ενίσχυση θεσμικών ε, οργάνων και αντιμετώπιση των κλιματικών απειλών και κατά πόσο λειτουργεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν πρέπει να αλλάξουμε την εστίασή μα. Είχαμε ένα πρόγραμμα δύο ημερών, συνεδριάσαμε με την Αντιπρόεδρο και με άλλα μέλη του, του Εθνικού Κογκρέσου, εκπροσώπου Τη της κυβέρνησης, ε, αρχές της Ονδούρας, ε, διεθνείς οργανώσεις ε, ανάπτυξης συνεργασίας για την ανάπτυξη και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις εργοζομένων, οργαδοτών και Πρέσβης των κρατών μελών. Και επίσης υπήρχε και μία επιτόπου επίσκεψη σε ένα πρόγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος FLEGT. Το βασικό πόρισμα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν πολύ σημαντικέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα, την ένδια, την ανισότητα, τη διαφθορά, τη βία, την γενικευμένη ατιμορρησία. Επίση, επισημάναμε ότι η κατάσταση στη χώρα έχει βελτιωθεί κάπω τα τελευταία χρόνια και τα προγράμματα για την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, χάρη κυρίω ε, στα όσα έκανε η ε, εκεί αντιπροσωπεία. Ε, παρά τι πρόσφατε μεταρρυθμίσεις υπάρχει εντύπωση ότι η διαφθορά και η ατιμορρησία εξακολουθούν να κυριαρχούν στη χώρα και αυτό φυσικά δεν επιτρέπει την βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πιο ευάλωτου, γυναίκες, μετανάστες, ε, ε αυτόχθονες πληθυσμούς, ε, δημοσιογράφους και άτομα που δραστηριοποιούνται στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι συνδυασμόν πολλών παραγόντων, αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, διακίνηση ναρκωτικών, εργασία των παιδιών και των εφήβων, ε, υπάρχει ατιμορρησία, γενικότερη διαφθορά και ε, πολύ μεγάλα ποσοστά ανισότητας. Να σας δώσω και κάποια στοιχεία τα οποία σας δείχνουν λίγο καλύτερα την πραγματικότητα. Καταρχάς, το ποσοστό δολοφονιών γυναικών είναι ε, επονίδιστο περίπου 40 γυναίκες το μήνα δολοφονούνται, που σημαίνει ότι κάθε μερικές ώρες έχουμε μία δολοφονία μιας γυναίκες. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, εγκυμοσύνες πριν από τα 25, πολλές εκ των οποίων είναι αποτέλεσμα βιασμού, που σημαίνει ότι το 12% των ανηλίκων γυναικών θα εγκυμονήσουν λόγω βιασμού. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο φέτος ε, δολοφονήθηκαν 42 φοιτητές, 5 ε, άτομα που εργάζονται στη δικαιοσύνη, 95 μεταφορείς, 45 ε, εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και 27 σε δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, σε 10 χρόνια πέθαναν περίπου 45.000 άτομα από δολοφονίες. Αυτό ε, σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί το ποσοστό της ατιμορρησίας που βάσει του παρατηρητηρίου υπερβαίνει το 70% των περιπτώσεων. Τμήμα της έλλειψης ασφάλειας προέρχεται και από την ίδια την αστυνομία, τη στρατιωτική αστυνομία ε, και ε, του ίδιου του στρατού που ορισμένε φορές είναι συνένοχος μαζί με το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροβόλα όπλα και νόμιμα και παράνομα και ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η νομοθεσία επιτρέπει να διαθέτει ο κάθε άνθρωπος μέχρι πέντε όπλα. Ε, οι ε, προασπιστές των ε, θεμάτων περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης και τα θέματα των ΛΟΑΔ, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές δολοφονίες που βρίσκονται ουσιαστικά στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, με ανήσυχε και το γεγονός ότι είχαμε σκηνές βίας και στα μέσα ενημέρωσης. Ε, αν το μέλλον μιας χώρας είναι τα παιδιά και η παιδεία, είναι ακατανόητο να δείχνουν ανα πάσα στιγμή της ημέρας τις συνθήκες δολοφονίας και μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο έχουν ε, βρεθεί δολοφονημένη. Ε, τα παιδιά ουσιαστικά ε, συνηθίζουν τη βία και τη θεωρούν λογική. Βλέπουν εικόνες οι οποίες είναι περισσότερο εικόνες ταινιών για κάποιους άλλους από την πραγματικότητα. Επίσης είναι σύνηθες τα μέσα επικοινωνίας να μην παρουσιάζουν απόλυτα την πραγματικότητα. Διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν οποιαδήποτε δήλωσή μας πριν πάμε και εγώ ως επικεφαλής αποστολής αποφάσισα να μην κάνω καμία δήλωση πουθενά για κανένα θέμα, σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Ακόμα και έτσι την επόμενη μέρα ε, μετά την άφηξή μας εμφανίστηκαν άρθρα στον τύπο που όπου ε, έλεγε ότι οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν την πρόοδο της κυβέρνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε ανοίξει το στόμα μας. Αυτό δείχνει απλώς πώς έχει κατάσταση στον τύπο ε, ορισμένες φορές υπάρχουν εντελώς διστάμενες απόψεις ε, με τους συνομιλητές μας όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική κατάσταση και αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη σύγχυση και αυτό επιδεινώθηκε γιατί βρισκόμασταν και σε προεκλογική περίοδο η οποία ήταν και με ιδιαίτερη ένταση. Ε, αυτό κυρίως φάνηκε σε θέματα όπως ποινικοποίηση των αμβλώσεων και κοινωνικές και εργασιακές ελευθερίες. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πιο ειλικρινής και πιο εύκολος πολιτικός διάλογος και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ονδόρα ακόμα δεν έχει εφαρμόσει καμία από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ε, ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές οργανώσεις ε, μας παρουσίασαν και την ανησυχία τους ε, την περίπτωση που επανεκλαγεί ο Πρόεδρος για την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων μετά την επανεκλογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι χορηγοί θα πρέπει να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο και να πιέζουν τι κυβερνήσεις για αυθεντική αλλαγή που θα περιλαμβάνει τους πάντες. Και φυσικά ε, υπάρχουν και εργασίε τη Νέα οικονομική και κοινωνική επιτροπή, η οποία συστήθηκε χάρη στο πρόγραμμα Eurosocial τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που διευκολύνει ε, λίγο τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, αλλά εκκρεμούν πάρα πολλά πράγματα. Πολλέ ε, πρόσφατες μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να μην είναι αποτελεσματικέ και άρα σημαίνει ότι δεν έχει γίνει πραγματική υλοποίηση στην πράξη. Ε, λόγω έλλειψη και ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών ε, πόρων και υποδομών. Ορισμένε φορέ διαπιστώθηκε ότι αυτό προέκυψε από έλλειψη πολιτικής βούλησης των αρχών της Ονδούρα. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι εκκρεμούν πάρα πολλά, η στήριξη στον προπολογισμό και οι δυνατότητες πολιτικού διαλόγου μαζί με τα προγράμματα ε, τεχνικής υποστήριξης ε, ε, ε, οδηγούν σε μια ικανοποιητική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονδούρας, ε, ιδίω στον τομέα της επιστημιστικής ασφάλειας, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την εργασία και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου έχουν επιτευχθεί κάποια σημαντικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η εξέλιξη μιας νομοθεσίας για τους δημοσιογράφους, ε, δικαστές, ε, ακτιβιστές ε, που έγινε με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία καταδεικνύει ότι ναι μεν υπάρχει η νομοθεσία στο χαρτί, δεν υπάρχει η βούληση να το υποστηρίξουν με κατάλληλο προϋπολογισμό όλα αυτά. Ε, μία θετική πτυχή είναι ότι υπάρχει στάση συνεργασίας της κυβέρνησης για το διεθνή έλεγχο. Ε, όπως για παράδειγμα η σύσταση ενός γραφείου της, ε, ε είπα, της εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, με την Όσον αφορά την εμπορική συμφωνία η οποία ε, τέθησε ισχύ μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης, είναι πολύ σημαντικό ε, να εγγυηθούν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει της Σύμβασης 169 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και να λάβουμε υπόψη μας τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα προγράμματα FLEGT είναι καλά για άλλους τομείς. Και για να ολοκληρώσω, η σύστασή μα είναι η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ονδούρα να συνεχίσει τι προσπάθειε για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, το κράτο δικαίου, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω στήριξη προπολογισμού και πολιτικού διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνάδελφε, και εμείς ευχαριστούμε για την αναλυτική και περιστατωμένη ανάλυση που μα κάνετε σχετικά με το ταξίδι σα στην Ονδούρα. Ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ενημερώσω την Επιτροπή ότι αυτού εξοχότητα ο πρέσβης της Ονδούρας ε, έστειλε επιστολή στην Επιτροπή και μας είπε ότι δυνατή σήμερα να παραστεί στην συνεδρίαση. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντελαριτσία, επικεφαλής της Μονάδας για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να μας κάνει τα δικά του σχόλια. Muchas gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Ντελαρίτσιο. Σας ευχαριστεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊκής ε, Δράσης για την ευκαιρία μας δίνεται να κάνουμε αυτή την παρουσίαση και επίσης είναι πάρα πολύ θετική η συνεργασία που έχει γίνει και πριν την ε, αποστολή και στην Τέγκουσικάλπα υπήρξε όλη η υποστήριξη που χρειάστηκε, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί είχαμε την αποχώρηση του προηγουμένου πρέσβεως και λοιπά. Και πάρα αυτά είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε την ε, αποστολή και να αποκτήσουμε μια πλήρη εποπτεία για το τι ισχύει στη χώρα. Η συνεργασία με τη χώρα είναι η πιο, δεύτερη πιο σημαντική για τη Λατινική Αμερική. πιο σημαντική. Και έτσι έχουμε και λειτουργία παρατήρησης, είχαμε επίσης και μια αποστολή του ηλεκτρικού συνεδρίου, οπότε και αναλύθηκαν τα σχετικά με την ε, συνεργασία με την χώρα και είχαμε και την αποστολή της Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ, πολύ σημαντικά στοιχεία για μας, γιατί από τις σχετικές εκθέσεις προκύπτει ότι γενικά η συνεργασία μας είναι σε επίπεδα ικανοποιητικά. Και πάντοτε βέβαια υπάρχει έδαφος για βελτίωση. Πάντοτε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια στη καθημερινή βάση και οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ πολύτιμα όλες αυτές οι εισηγήσει για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Όντως έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας και τέτοιου είδους εκθέσεις για μας αποτελούν ένα κίνητρο και να βελτιώσουμε έτσι τις επιδόσεις μας στη συνεργασία, να βελτιώσουμε τον πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση. Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής έναντι της χώρας ε, είπαμε ότι βέβαια η υπόθεση τη προστασία των δικαιωμάτων είναι κάτι το εγκάρσιο, κάτι το οριζόντιο για όλα τα θέματα τη συνεργασία μα, γενικά για την ε, ευρωπαϊκή παρουσία εκεί. Κομβικό θέμα, κεντρικό όσον αφορά τη συνεργασία. Και έχουμε επίσης τις πιο χτυπητέ περιπτώσεις, όπως η υπόθεση που αναφέρατε, η υπόθεση Κάθερες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δραστήρια. Συμμετέσχε και στις δικαστικές νομικές εξελίξεις. Έχουμε επίσης και τους ε, εσωτερικά εκτοπισμένους. Έχουμε τα θέματα τα σχετικά με τα δάση. Και ήταν πολύ χρήσιμο και για εσάς το ότι επιτόπου πήγατε και δείτε τι γίνεται με το πρόγραμμα FLECT. και σύντομα πρόκειται να ολοκληρώσουμε τη σύνευση της συμφωνίας και το πιο σημαντικό είναι να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι εμπορική συμφωνία. Βέβαια το αρχικό TAF στο FLEGD σημαίνει trade, εμπόριο, αλλά να το θεωρήσουμε αυτό είναι ένα εργαλείο, ένα εργαλείο για να έχουμε μια πιο άρτια διακυβέρνηση. Γιατί σε μια τέτοια χώρα έχουμε και επαρχίες όπου κατοικούν οι θαγενείς, οι ντόπιοι και επομένως εκεί ρίχνουμε το βάρος μας και εκεί προσπαθούμε να έχουμε μια πρώτερη ε, διαβούλευση με αυτούς τους ε, ανθρώπους, τους ηθαγενείς και να γίνεται έτσι η σχετική ενημέρωση όσον αφορά και τα όσα προβλέπουν οι διεθνείς συμφωνίες εργασίας. Άρα, θα βοηθήσει αυτή η συμφωνία θα είναι θετικό βήμα. Ελπίζουμε να λυθούν κάποια εκκρεμούντα προβλήματα. Ε, επίσης, να σας ε, ευχαριστήσω και να σας διαβιώσω ότι η έκθεσή σας για μας είναι κίνητρο για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντελαρίτσια και τώρα θα μου, δώσετε, την ευκαιρία να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπέρδο από τη Γενική Διεύθυνση για την Αναπτυξιακή Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπέρδο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μούτσα ε, gracias, σενιόρα πρεσίδεντα, Και εγώ να συνεχίσω να σας τα πω στα αγγλικά, μια που όλο ισπανικά ακούγονται. Μητρική μου γλώσσα να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης. Άλλη μια φορά. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Και με την κυρία Σάντζεθ και με τους συναδέλφους. Ε, βέβαια και είμαστε άκρος ικανοποιημένοι που αυτή η έκθεση αναφέρει ότι ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας της υπηρεσίας μας βοήθησε για τις βελτιώσεις που είδε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αναβίβολο επίση. Συμφωνούμε και με το άλλο σημαντικό. Την σύνεψη που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε αυτή τη συμφωνία με τη χώρα για που έχουμε κάποιες ε, προκλήσεις, κάποια προβλήματα πολύ σημαντικά για διάφορους τομείς. τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι οριζόντια θέματα τα οποία μας απασχολούν για όλα τα προγράμματα τα οποία τρέχουμε. Επίσης, ο ρυθμός διαμόρφωσης προγραμμάτων στους τρεις Τομεί που αφορά η δράση μας με πολυμερή χαρακτήρα, η διατροφική ασφάλεια, επασχόλησε και το κράτος δικαίου δηλαδή. Οπότε είπαμε ότι τα διαπερνούν αυτά τα προγράμματα, αυτά τα ζητήματα, διαφθορά, ανθρώπινα δικαιώματα που τα προσέχουμε πάρα πολύ. Να μην υπησέλθουμε τώρα στις λεπτομέρειες για κάθε ένα πρόγραμμα από αυτά τα οποία μπορέσαμε να τρέξουμε από το 2014. Πάντως σήμερα υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας και το τονίζω ακριβώς όπως ε, είπε και ο κ. Ντελερέτσι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει και τεχνικός, τεχνοκρατικός διάλογος και πολιτικός με τους διάφορους τομείς αλλά και με τις ε, αρχές της χώρας αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Διάλογος ο οποίος είναι πολύ καλύτερα δομημένος, είναι πολύ πιο ζωντανός από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Ε, έτσι πάμε προς το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή νέα νομοθεσία στους τομεί για τους οποίους συνηθιζόμαστε και επίσης χάραξη κάποιων πολιτικών. Πολύ σημαντικό όλα αυτά. Τώρα ήρθε η ώρα, όπως είπε η κυρία Σάντσεφ, να παρακολουθήσουμε το πώς θα εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, πώς θα ασκηθούν οι σχετικές πολιτικές. Να, τα είπαμε για την πολιτική απασχόληση που θα μπορούσε να βοηθήσει την ε, χώρα και να υπάρξει δυναμική πολιτική στο μέτωπο της απασχόλησης και να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί για τους στόχους που έχουν τεθεί για την περίοδο μέχρι το 20. Επίσης θα πρέπει να επενέσουμε πέραν των ε, προγραμμάτων, τη δημοσιονομική βοήθεια που παρέχεται ε, για τα δασικά. Διατροφική ασφάλεια επίσης. Έχουμε και κάποια άλλα ελάσσονα προγράμματα Φερρυπίν με το εργαλείο για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά πιο μικρά είναι από πλευρά Όμως αυτά μπορούν που ουσιαστικά να βοηθήσουν τους δικαιούχους όπου εφαρμόζονται. Πάμε πιο μικρά έργα και προγράμματα τα οποία καλύπτονται από αυτό το εργαλείο δημοκρατίας και δικαιωμάτων και επίσης έχουμε το project το οποίο χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαχειριζόμαστε εμείς και αφορά ανηλίκους και εφήγους. Για να το μεταφράσω, τους εξαναγκαστικά η βία εκτοπιστέντες. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιδόσεις αυτές και τη χρηματοδότηση σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκατοντάδες νέων και παιδιών που βρίσκονται σε τέτοια ευάλωτη θέση. Εδώ να βάλω μια τελεία, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση, για αυτή την παρουσίαση. Πρόεδρος. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Μπέρκο και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, συναδέλφους αν έχουν κάποιες ερωτήσεις ή αν θέλουν να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένα συνάδελφος, ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω απλώς ότι προφανώς και είναι τραγικό να χάνονται αυτές οι ζωές. Ε, ε, ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ονδούρα και το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, το οποίο συζητούμε συνεχώς. Έχω εδώ ένα φυλάδιο για τα όσα έκανε ο πρόεδρος Ερνάντες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά στην ουσία είναι ε, μία, ένας εξοραϊσμός της πραγματικότητας της Ονδούρας. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών στην Ονδούρα, το οποίο πολύ σωστά ετέθη ε, από τους προλαλήσαντες. Και το Πανεπιστήμιο της Ονδούρας είπε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2017 δολοφονήθηκαν 177 γυναίκες και μιλάμε για το πρώτο εξάμεινο. Κάθε 18 ώρες έχουμε μια δολοφονία μιας γυναίκας. Και αυτό το φυλάδιο είναι πάρα πολύ ωραίο, εικονογράφηση, και ουσιαστικά είναι απλώς ε, το εγκόμιο του καθεστώτος. Δεν γράφει όμως τίποτα για την πραγματικότητα της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τελαρίτσια για αυτά που είπε. Ε, όπως είπε πολύ σωστά, εκκρεμούν ακόμα πάρα πολλά και είναι καθήκον μας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθήσουμε από κοντά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αρχές της Ονδούρας να εφαρμόσουν ε, γενικές πολιτικές ε, οι οποίες θα συνάδουν με μια σύγχρονη χώρα η οποία θέλει να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρότασή μου λοιπόν κυρία Πρόεδρε είναι για του χρόνου. Δυστυχώς εγώ φέτος δεν μπορούσα να ε, μεταβώ με την αντιπροσωπεία στην Ονδούρα και ήταν εξαιρετική η ιδέα της αντιπροσωπείας μας ε, να πάει και να στείλει μέλη για να δουν επιτόπου την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε και του χρόνου και να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, να δούμε τι γίνεται με τις εξελίξεις ε, τα επόμενα χρόνια, να δούμε αν οι αρχές της Ονδούρας ε, θα μπορέσουν να έχουν κάποια πρόοδο. Να ευχαριστήσω και την κυρία Σάντσε για την ε, έκθεσή τη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ε, ξέφρασε πάρα πολύ εύγλωτα την κατάσταση στην Ονδούρα και καθόρισε, μας παρουσίασε τα προβλήματα σαφέστατα. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Φαρία. Ήταν πολύ σημαντικέ οι επισημάνσει που κάνατε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο να τοποθετηθεί. Τότε θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο και μια ερώτηση, να απευθύνω μια ερώτηση. Ε, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και εγώ στο επικοδομητικό έργο της, ε, που παράγει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ονδούρα. Το έχουμε πει και στις άλλες προηγούμενες συνεδριάσεις των επιτροπών μας. Έργο που είχαμε την ευκαιρία, όπως είπαμε και προηγουμένως, να αξιολογήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών της για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, της κοινωνικής συνοχής, της αηφόρα ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζεται και δημιουργεί μια θετική εικόνα για την ε, αντιπροσωπεία μας εκεί. Ε, είπατε κυρία Σάντζεθ, ότι η χαόδης κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση που εμφανίζει η χώρα με την ανισοκατανομή της διανομής του πλούτου και της ιδιοκτησίας αντανακλάται σε όλες τις δομές του κράτους δημιουργώντας φαινόμενα διαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας. Μα είπατε ότι η αντιπροσωπεία τη ΔΕΒΕ διαπίστωσε ότι πολλέ πρόσφατε νομικέ μεταρρυθμίσει παραμένουν αναποτελεσματικέ εξαιτία τη αναποτελεσματική εφαρμογή και τη έλλειψη ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων αλλά και των υποδομών του. Επίση, στην έκθεση σημειώνεται ότι σε ορισμένε περιπτώσει διαπιστώθηκε έλλειψη πολιτική βούληση ω προ αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρακαλέσω να μα ενημερώσετε πιο συγκεκριμένα και να ρωτήσω και τον κύριο Ντελαρίτσια από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αν θα ήθελε να σχολιάσει ή αν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Θα απαντήσετε εσείς. Ναι, με συγχωρείτε. Όσον αφορά την πολιτική βούληση, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Υπήρχε όμως ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε και θα μπορούσα να σας δώσω ως παράδειγμα. Είχαμε συνάντηση με την Υπουργό Αρμόδια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη ρωτήσαμε για αυτό το νόμο ε, και όντως ο νόμος γιατί ο συνήγορο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ καλός, είναι εξαιρετική δουλειά και λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν και η υπουργό, όταν τη ρωτήσαμε τι γίνεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας, πώς προχωράει, ε, τι έχουν προβλέψει στον προπολογισμό, αν υπάρχουν κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι, τεχνικοί πόροι, υποδομές κλπ. Μας είπαν ναι, Βεβαίως ε, έχει συστηθεί ένα γραφείο εδώ στο γραφείο του Συνηγόρου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάρα πολύ μεγάλο γραφείο, πολύ κόσμο, ε, πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και την επόμενη μέρα συναντήσαμε το διευθυντή του γραφείου και ο διευθυντής ε, του γραφείου διέψευσε όλα όσα μας είπε και μας είπε ότι δεν τους και το προσωπικό, είναι πάρα πολύ λίγο ο κόσμο. υπάρχουν ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, ελάχιστοι τεχνικοί πόροι, δεν έχουν εμπειρογνώμονε, ε, πρέπει να ε, προσληφθούν περισσότερα άτομα και να υπάρχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο γραφείο. Αυτό είναι αυτό το οποίο μα εντυπωσίαζε. Ανάλογα με το ποιον μιλούσαμε, ποιον συναντούσαμε, ακόμα και άνθρωποι που εργάζονται για την κυβέρνηση, σου παρουσιάζουν τελείω διαφορετική εικόνα για το ίδιο θέμα. Και το ίδιο γεγονός που μας οδηγεί και στην εντύπωση ότι ούτε καν αυτοί οι ίδιοι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εδώ στο γραφείο για την ε, προάσπιση των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουν ενδιαφερθεί ιδιαίτερα. Ο υπουργό μας λέει με ένα πράγμα και μετά ο διευθυντής του γραφείου μας λέει εντελώ το αντίθετο, σε λιγότερο από 24 ώρες, ε, ε, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι απλώς ε, παράδειγμα το οποίο εξηγεί αυτό που διαπιστώσαμε, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει το σύστημα. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας. Μας εξήγησε το πρόγραμμα Ονδούρα 2020, πράγματα που περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο είναι η προώθηση και η διεύρυνση των ε, ε, ε δυνατότητων κλωστοφαντουργίας και θέλουν να μπουν και στην αγορά. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση έχει ένα όραμα ανάπτυξης της χώρας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είναι αυτές οι θέσεις εργασίας που θα οδηγήσουν σε κατάρτιση κόσμου και δεν θα υπάρξει ψηλή και τον ρώτησα κατά πόσον θεωρεί ότι στη χώρα του ε, υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερες δουλειές από το να ε, ράβει για 18 ώρες ε, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αυτά τα επαγγέλματα αλλά είναι μια χώρα που από ό,τι φαίνεται επικεντρώνει στην παραγωγή της στην εξαγωγή υπηρεσιών πολύ μικρής προστιθέμενης αξίας και επομένω μου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στο λαό τη ε, και δεν έχει καμία ελπίδα ότι ο λαό θα μπορούσε να παράγει καλύτερα πράγματα με βοήθεια και στην εκπαίδευση κλπ. κλπ. Κάτι άλλο το οποίο μα εξέπλεξε είναι ότι ο Υπουργό μα είπε ότι υπάρχει περίπου ένα 30% ε, θέσεων στο σχολείο για όλους τους σπουδαστές που θα έπρεπε να έχουν τα σχολεία. Και ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυσης για να ανοίξουν περισσότερα σχολεία, να υπάρχουν περισσότερες θέσεις στα σχολεία για τα παιδιά, διότι αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι το 70% των παιδιών ε, στην Ονδούρα δεν έχουν σχολείο να τα στεγάσει και δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στο σχολείο. Ε, Αυτά είναι θέματα πολιτική βούληση, όπω σα έλεγα. Επομένω για αυτούς, αυτά φάνηκαν ότι είναι θέματα ίσονα σημασία. Η παιδεία, δηλαδή, φαίνεται ότι δεν του ενδιαφέρει και πάρα πολύ, διότι θέλουν φθηνά εργατικά χέρια, σε συνθήκε σχεδόν σκλαβιά. Επομένω και όλα έρχονται εκεί να, βρεθούν στο σωστό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντελαρίτσια. Ε, Κύριε Πρόεδρε, να το αναλύσουμε στο πλαίσιο της ιστορίας της χώρας, μια που η πανεπιστημιακή θεωρούν ότι αυτό είναι καπιταλιστικό σύστημα, πρότυπο ανάπτυξης. Κάτι το οποίο διατρέχει όλη την ιστορία της χώρας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει η πρόθεση του να προσδώσουν κάποιο χαρακτήρα, κάποιο ένδυμα νομιμοποίηση για αυτού του στόχου. Έχουμε αυτό το νόμο της προστασία των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φερρυπίν. Επίσης ο, ο νόμος χρηματοδότησης των ε, κομμάτων ε, που υποστηρίχθηκε από Ματσί και από εμά. Επομένω πρόκειται για αυτή την νομοθεσία, του σχετικούς ε, πόρου. οι χωρί τους πόρους είναι νεκρογράμμα η νομοθεσία, άρα και εμεί θα πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και στα πλαίσια ενό ανοιχτού και ειλικρινού διαλόγου να φροντίσουμε αυτές οι πρωτοβουλίε να βελτιώσουν την κατάσταση. Και να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικές αυτές οι ιδέες. Είναι φυσικά πολύ σημαντική υπόθεση η παιδεία και εκεί συνεργαζόμαστε για να δούμε πώς μέσα από τις επαφές μας με την κυβέρνηση, με το διάλογο, τη συνεργασία, θα βοηθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Αφετηρία μας και το πνεύμα μας είναι ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποιο σχόλιο ή να πάμε στο επόμενο σημείο. Προχωράμε. Στο σημείο 5 λοιπόν που αφορά στην πολιτική κατάσταση στη Γουατεμάλα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια συνοπτική αναφορά, θα σας κουράσω λίγο, για τα περιστατικά που σηματοδότησαν την τελευταία πολιτική κρίση στη Γουατεμάλα. Στις 27 Αυγούστου του 2017, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γουατεμάλα, κύριος Μοράλες, ανακήρυξε τον κύριο Βελάσκες, επίτροπο της Διεθνούς Επιτροπής κατά της ατιμορρησίας στη Γουατεμάλα, ως persona non grata και διέταξε την απέλασή του από τη χώρα. Η Διεθνής Επιτροπή κατά της ατιμορρησίας που βρίσκεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη συνεχιζόμενη διαδικασία πρόθεση των μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης των κρατικών θεσμών καθώς και στην αποκάλυψη πολυάριθμων σκαντάλων διαφθοράς στην Γουατεμάλα. Από το 2007 μέχρι και σήμερα η ΣΥΣΥΚ έχει διενεργήσει περισσότερες από 200 έρευνες, εκ των οποίων οι περισσότερες από τις 160 έχουν οδηγήσει σε απαγγελίες κατηγοριών εναντίον προέδρων, υπουργών, πρώην διευθυντών της Εθνικής Αστυνομίας, απόστρατων στρατηγών, πολιτικών, επιχειρηματιών, εμπόρων ναρκωτικών, εκτελεστών κλπ. Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η αντιπροσωπεία μας έχει επανειλημμένα στηρίξει το έργο και την εντολή της ΕΣΥΚ για τον λόγο αυτό, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κεντρική Αμερική εξέδωσε δήλωση που υπεγράφει από εμένα με την ιδιότητα της Προέδρου και τους δύο αντιπροέδρους σχετικά με την απέλευση του Επιτρόπου Βελάσκετ από την Γουατεμάλα, η οποία και έχει περιληφθεί στο φάκελό σας που σας έχει ήδη διανεμηθεί. Δύο μέρες πριν από την ανακοίνωση του Πρόεδρου κ. Μοράλες, ο κ. Βελάσκετ και η κυρία Αντάντα, Γενικός Εισαγγελέας, είχε ζητήσει από το Συνταγματικό Δικαστήριο την άρση της πολιτικής ασυλίας του κυρίου Μοράλες προκειμένου να προβεί στην απαγγελία κατηγοριών που συνδέονται με παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας. Η απόφαση του Προέδρου να πελάσει τον Επίτροπο Βελάσκες ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο και ο Επίτροπος παρέμεινε στη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με του σχεσμού τη Γενική Εισαγγελία, το Εθνικό Μέτωπο Σύγκληση, που είναι το κόμμα του κ. Μοράλε, δεν δήλωσε το ποσό των 6,7 εκατομμυρίων κετσάλ, περίπου 780.000 ευρώ που προερχόταν από εισφορέ στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Μόράλε το 2015 στο Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο, όπω απαιτείται από τον εκλογικό νόμο. Ο κ. Μοράλε που είχε στυλιτεύσει ω υποψήφιο πρόεδρο πρακτικέ αυτέ, είχε κατά επανάληψη αρνηθεί τι κατηγορίε. Παρ' όλα αυτά, στι 11 Σεπτεμβρίου του 2017, το Κογκρέσο τη Γουατεμάλα απέρριψε την αίτηση άρσης ασυλία του Προέδρου Μοράλε. Και επιπλέον, το Κογκρέσο ενέκρινε δύο, μετα... δύο μεταρρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, για τις οποίες ασκείται σκληρή κριτική, καθώς φαίνεται ότι λειτουργούν προς όφελος των κομματικών ηγετών με στόχο την προστασία τους από καταγγελίες για την παραβίαση των κανόνων χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατιών. Το Συνταγματικό Δικαστήριο και πάλι υποχρέωσε το Κογκρέσο να υπαναχωρήσει, με το αιτιολογικό ότι καθότι εν λόγω τροποποιήσει οδηγούν στην καταστρατήγηση των κανόνων χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών και επιτρέπουν σε ορισμένου εγκληματίε που εκτείουν ποινέ κάτω των 10 ετών να αφήνονται ελεύθεροι με αντάλλαγμα ένα μικρό πρόστιμο, υπονομεύουν το κράτο δικαίου. Αυτέ οι ενέργειε του Πρόεδρου Μοράλε και του Κογκρέσου προκάλεσαν τι αντιδράσει δεκάδων χιλιάδων πολιτών στη Γουατεμάλα οι οποίοι στις 20 Σεπτεμβρίου διαμαρτυρήθηκαν διαδηλώνοντας, θυμίζοντας τις μεγάλες διαδηλώσεις που προηγήθηκαν της παρέτησης του πρώην Προέδρου κ. Πέρες Μολίνα. Ο κ. Μοράλης είχε ταχθεί υπέρ της ΣΥΚ, όταν αυτός ανέλαβε την εξουσία και μάλιστα ήταν αυτός που ανανέωσε για πέμπτη συνεχή φορά την εντολή της στις 16 Απριλίου του 2016. Ωστόσο, τον Αύγουστο κατηγόρησε τον επικεφαλής ερευνητή κ. Βελάσκετ ότι υπερβαίνει την εντολή συμμετέχοντας ο ίδιος σε, εσωτερικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην ευθύνη του κράτους της Γουατεμάλας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ΔΕΚΑΜ επισκέφθηκε τη Γουατεμάλα από 16 έως και 18 Φεβρουαρίου του 2015 και ότι με την ευκαιρία αυτή είχε μακρά και ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Γενική Εισαγγελέα κυρία Αλτάνα γενική εκτίμηση που αποκομίσαμε τότε σαν αντιπροσωπεία είναι ότι η κυρία Αλντάνα επιτελεί ουσιαστικό και σημαντικό έργο και ελπίζουμε να συνεχίσει το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει και να υποστηριχθεί με κάθε δυνατό τρόπο από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Μοράλες εξήγηλε την πρόθεσή του να αναθεωρήσει την Ιδρυτική Συμφωνία της ΕΣΥΚ. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι παρέλαβα δήλωση με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου του 2017 από την Πρεσβεία της Γουατεμάλα, στην οποία η κυβέρνηση της Γουατεμάλα παρουσιάζει τη θέση της σχετικά με τη ΣΥΣΥΚ. Η επιστολή αυτή επισυνάπτεται στο φάκελό σας. Επιπλέον, να σας ενημερώσω ότι η αυτού εξοχότητα ο κύριος Γκουτιέρετ, πρέσβης της Γουατεμάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πληροφόρησε ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την πληροφόρηση και θα μου επιτρέψετε να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντελαρίτσια, προϊστάμενο τη Διεύθυνση για την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και την Καραβική τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Κύριε Ντελαρίτσια, έχετε το λόγο. Κύριε Ντελαρίτσια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί από κοντά τι πρόσφατε εξελίξει στη χώρα και ανησυχούμε βαθύτατα με αυτές τις ε, απόπειρες φραγμού ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είμαστε ιστορικός εταίρος και πιστά βοηθάμε τη χώρα να καταλμίσει την διαφθορά. Και βοηθά βέβαια πάρα πολύ αυτή η Επιτροπή Καταπολέμησης της ε, Διαφθοράς σε στενή συνεργασία με την Γενική Εισαγγελία. Ακριβώς όπως τονίστηκε από τον εκπρόσωπό μας στις 28 Αυγούστου, το έργο της ε, Γενικής ε, Εισαγγελίας και της Επιτροπής για την Καρβούνωση της Ατιμορρησίας ήταν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στην καταπολέμηση ατιμορρησίας και διαφθοράς. Αυτά τονίστηκαν στη 16 η έκθεση της Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε και εκεί αποτυπώνονται όλες οι επιτυχίες που έχουμε καταφέρει. Όλα αυτά που η Επιτροπή κατάφερε σε συνεργασία με την Εισαγγελία. Και όλα αυτά ελπίζουμε ότι με αντικειμενικό τρόπο θα τα ζυγίσουν, θα τα λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιες ε, άρχες. Και στις δηλώσεις μας τονίζουμε πόσο σημαντική κάνει αυτά τα δύο θεσμικά όργανα στην υπόθεση του κυρίου Βελάσκεθ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν παρεμβάσεις στο έργο αυτών των φορέων. Εμεί συνεχίζουμε πιστά να υποστηρίζουμε τον αγώνα της χώρας κατά διαφθοράς και ατιμορρησίας και πέρα του κράτους δικαίου. Αυτές οι προσπάθειες είναι απαραίτητε και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και γενικότερα, ούτως ώστε να υπάρξει ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, κάτι το οποίο θα ωφελήσει το λαό της χώρας. Ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση. Να κύριε Φαρία. Πρώτα, πρώτα, κυρία Πρόεδρε, για άλλη μια φορά να συγχαρώ μια που έγιναν αυτά τα διαβήματα και που στους φιναλίστ και τέλος πάντων ψήφου για το βραβείο Ζαχάροφ προτείνεται και αυτή την κυρία. Μπορούμε να πούμε ότι η διαφθορά και η φτώχεια στη χώρα είναι ένας φαύλος κύκλος που συνεχίζεται. Έχουμε επίσης παράνομη χρηματοδότηση σε προεκλογικές εκστρατείες. Μπλέκεται εκεί και ο πρόεδρος Μοράλες. Ήθελε να πελάσει τον Επίτροπο και όπως σωστά μας τα είπατε κυρία Πρόεδρε. Χρησιμοποιεί ό,τι μέσα μπορεί και μέσα στο Κογκρέσο, στην Εθνοσυνέλευση τέλο πάντων και σε όλους τους χώρους, σε όλα τα βήματα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο λαός της χώρας δεν έχει κράτος. Το έργο της αντιπροσωπείας μας, όπως και εσείς εξηγήσατε, είναι να δούμε πώς θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Γενικότερα στην Κεντρική Αμερική. Πάντως για την περίπτωση της Γουατεμάλας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως εάν η Γουατεμάλα συνεχίζει να καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει κάτι να κάνουμε, θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα στη χώρα ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και Μπορούμε να αναλάβουμε δράση με πολλούς τρόπους. Έχουν πολλά μέσα στη διάθεσή μας, όπως τα ξέρετε καλύτερα από μένα, Πρόεδρε. Κρίμα που δεν ήρθε ο προσβευτής εδώ. Αλλά πώς να καταπολεμηθεί η διαφθορά ε, όταν δεν το βλέπει στην καθημερινή ζωή ο λαός της χώρας. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το λαό της χώρας εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να συντάξουμε μία επιστολή με συστάσεις, με προτάσεις. Να απευθύνουμε την επιστολή στην κυβέρνηση της χώρας και να ζητούμε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να μην φαινόμενα σαν την απέλαση του κυρίου Βελάσκες, σαν την απόπειρα πέλας τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρία. Θα λάβουμε πολύ σοβαρά τις επισημάνσεις, θα τις ξανασυζητήσουμε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση, αν έχετε κάποιο άλλο θέμα να συζητήσουμε σημερινή συνεδρίαση. Εάν δεν υπάρχει, εγώ δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους εκλεπτούς ε, καλεσμένους μας, να, να σας ευχαριστήσω όλους για την σημερινή παρουσία σα. εδώ, να ευχαριστήσω τους διερμηνείς μας για την διερμηνία που μας παρήσχαν. Και θα ήθελα να πω ότι η επόμενη συνάντηση της αντιπροσωπείας μας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου του 2017 στις Βρυξέλλες. Ε, και θέλω να ενημερώσω από τώρα τα μέλη ότι η πρόθεση της ε, Προεδρίας είναι να οργανώσει μια εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων που θα εστιάζει στην δυναμική και στις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές εν ώψη της εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.